Μετά τον διορισμό του κυρίου Ιαν Ντάνκαν ε, ως μέλος ε, του Βρετανικού Κοινοβουλίου ε, χειρεύει η θέση του από τις 23 Ιουνίου. Επίσης η κυρία Κομοντίνη Κατσία αναλαμβάνει θέση στην, στο Μαλτέζικο Κοινοβούλιο και γι' αυτό χειρεύει η θέση της από τις 24 Ιουνίου 2017. Το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Νεγκρέσκου, ο οποίος ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και συνεπώς η θέση του χειρεύει από τις 30 Ιουνίου 2017. Ο κύριος ε, Τζον Φλακ ε, έχει αναλάβει θέση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και γι' αυτό οι κύριοι Μάθιους και Καν από τις 29 Ιουνίου 2017 αναλαμβάνουν την θέση αυτή, καθώς και ο κύριος Τζον Χόουαρθ από τις 30 Ιουνίου 2017, αντικαθιστώντας ε, αντιστοίχως την κυρία Φόρτ